Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, γαλλόφωνους ε, φίλους μου γιατί τα γαλλικά είναι πολύ πιο ε, εκτεταμένη γλώσσα. Τα αγγλικά είναι πολύ πιο σύντομα και έχω μόνο 15 λεπτά για να σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα 5 ετών. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε άλλη γλώσσα πλην των αγγλικών. Σε τελικά σχεδόν αδύνατο. Θεωρώ λοιπόν ή θέλω να ελπίζω ότι θα μου κάνετε πολλές ερωτήσεις ε, για να μπω σε διάφορα θέματα. Ξεκινάω με τα εξή. Όπως είπατε πρόεδρε, ζούμε σε χαλεπούς καιρούς. Ιδιαίτερα χαλεπούς καιρού. Γύρω μας βλέπουμε στο κουμπάνι ε, 3.600 θύματα στην Ουκρανία, περίπου ο ίδιος ε, αριθμός ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα από τον ιό έμπολα. Αν στρέψουμε το βλέμμα προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, στη Λαμπεντούζα, όπου, την οποία επισκέφτηκα πριν από λίγες μόνο ημέρες, και αν δούμε και τα ε, θέματα διεθνούς πολιτικής που μοιάζουν να είναι μακριά, δεν είναι έτσι, γιατί επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών μας. Θεωρώ λοιπόν ότι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι κάτι που μας ρωτούν οι πολίτες μας.

σε αυτό το δύσκολο καιρό, στους χαλεπούς όπως σας είπα καιρούς, τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εκπροσωπεί, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχουμε βέβαια εργαλεία στα χέρια μας, κυρίως μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε μια εξωτερική υπηρεσία και τα επόμενα πέντε χρόνια οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή πολιτική, ένα κοινό όραμα και μια κοινή στρατηγική. Και αυτό είναι το πρώτο μου καθήκον για τα επόμενα πέντε έτη να, ε, να φτιάξουμε μια πραγματική εξωτερική πολιτική. Ίσως ε, για κάποιους από εσά, δεν ξέρω, αυτό να έχει λίγο αφελές. Οι πολίτες λένε, μα έτσι κι αλλιώς ε, τα κράτη πάντα έχουν εξωτερική πολιτική. Κάποιοι άλλοι λένε, δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα 21η εξωτερική πολιτική. Και συμφωνώ μαζί τους. Παράλληλα όμως όλοι μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη εποχή και το δύσκολο κόσμο εάν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τις ευθύνες μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε σε μεγάλη κλίμακα και να αντιδρούμε από κοινού. Ένα μεγαλοπρεπές όραμα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να διαχειριστούμε την εποχή μετά την κρίση μεγαλοπρεπή και μεγαλόπουνα προγράμματα για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά όλα είναι προς το συμφέρον μας. Δεν υπάρχει ούτε μία εσωτερική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην συνδέεται με την εξωτερική διάσταση. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που σήμερα δεν μπορεί να τα κάνει μόνο του κανένα κράτος μέλος. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον μας να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Γιούγκερ στην ομιλία του τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή να κάνουμε πλήρη χρήση, να εξαντλήσουμε πλήρως το δυναμικό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε τώρα τι χρειαζόμαστε κατά την άποψή μου. Τρία πράγματα. Καταρχήν, χρειαζόμαστε μια μορφή ιδιοκτησίας εισαγωγικά σε όλα τα κράτη-μέλη, το όραμα να είναι κοινό από την αρχή. Είναι πολύ αργά όταν φτάνουμε απλά στο πώς θα συντάξουμε ένα κείμενο. Είναι πολύ αργά να αντιδρούμε με ένα τέτοιο τρόπο σε κρίση. Από την αρχή χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα. Γι' αυτό λοιπόν ε, τους πρώτους μήνες όταν θα αναλάβω το αξίωμά μου θα επισκεφτώ τις 28 πρωτεύουσες ξεκινώντας με την επόμενη Προεδρία, τη Λετωνία και θα συναντηθώ όχι μόνο με την κυβέρνηση και τους υπουργούς εξωτερικών, αλλά και με τα κοινοβούλια των κρατών μελών, με τους βουλευτές, αλλά και με ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, ε, δεξαμενές σκέψεις, ακαδημαϊκούς, με όλους αυτούς, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό για να σφυριλατήσουμε ένα κοινό όραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική. Να αρχίσουμε να το σφυριλατούμε. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι έχουμε πέντε χρόνια που θα τα περάσουμε μαζί. Το δεύτερο που θέλω να πω, θα είμαι ευτυχής εάν μετά από πέντε χρόνια δεν θα ε, λέμε εμείς και οι άλλοι όταν θα αναφερόμαστε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα αναφερόμεθα σε εμάς. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούν σε επίπεδο θεσμικό και γνωρίζω βέβαια ότι από αυτού φέρω ιδιαίτερη ευθύνη γιατί έχω πολλά καπέλα, πάλι σε εισαγωγικά, πολλές ιδιότητες, μπορούμε να τα παριθμίσουμε αν θέλετε. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε η δομή που υπάρχει να είναι αποτελεσματική, να υπάρχει συνεργασία. Δεν θα το ζητούσα αυτό, βεβαίως, εάν δεν ήμουν και εγώ πρόθυμη για συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα και ανακοίνωσα από την πρώτη μέρα που προτάθηκα ότι θα ε, μετακινηθώ με το γραφείο μου στο Μπερλεμό, που δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όχι, απλά θα εργαστώ έτσι ώστε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να είναι ο πυρήνας όλων των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς έτσι πρέπει να είναι. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα συγκαλώ συνεδριάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να μοιραζόμαστε τη δουλειά. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να συντονίζουμε όλες τις δράσεις που έχουν εξωτερικές προεκτάσεις με τους επιτρόπους εξωτερικών σχέσεων αλλά και με άλλους. Γιατί δεν υπάρχει κανένα χαρτοφυλάκιο που να μην έχει τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής. Και θέλω να αφαιρθώ κυρίως στην ενέργεια, στο περιβάλλον και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο κύριο Γιούνκα ότι... Συντονίσω και θα προεδρεύσω μια ομάδα που θα συνεδριάζει μία φορά το μήνα υπό διάφορου σχηματισμού ανάλογα με την ατζέντα και η πρώτη συνεδρίαση αυτή τη ομάδα θα γίνει την πρώτη εβδομάδα που θα αναλάβουμε τα καθήκοντά μα, αρχέ Νοεμβρίου. Επίση, μια και χρειάζεται να συντονιζόμαστε περισσότερο και πιο αποτελεσματικά εσωτερικά τι εσωτερικέ πολιτικέ και τι εξωτερικέ πολιτικέ υπάρχει αυτή η ομάδα. Αν δούμε τι βασικέ απειλέ και τι βασικέ προκλήσει για την ασφάλεια, χρειαζόμαστε αυτή, αυτό το συντονισμό. Τρομοκρατία. Μεταναστευτικέ ροέ ασφάλεια και άμυνα. Πρέπει να δουλέψουμε υπό διάφορους σχηματισμούς ανάλογα με τα θέματα. Ανέφερα την ασφάλεια και την άμυνα. Να σα πω λοιπόν ότι βασίζομαι στη μικρή, αλλά υπάρχουσα εμπειρία που έχω στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, αλλά και, στην, και στο ΝΑΤΟ και θεωρώ ότι η συνεργασία για αυτά τα θέματα Όπω προβλέπεται από τη στρατηγική ατζέντα που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο, μία από τι τέσσερι προτεραιότητας, άρθρο 21 τη συνθήκη, θα πρέπει να προχωρήσει. Θα πρέπει να εμποδίσουμε του πολέμου, να προωθήσουμε την ε, ειρήνη και να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία. Αυτό θα είναι ο με καθοδηγεί. Και μια και μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή είναι μια από τι ιδιότητέ μου, από τα καθήκοντά μου ω ε, επικεφαλή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα συνεργαστώ λοιπόν. Θα προεδρεύσω στα Συμβούλια Ασφάλειας και θα επισκεφτώ τις αποστολές μας. Βασίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας κυρίως για να βασιστούμε στην εμπειρία σας, στο όραμά σας, για να τα καταφέρουμε. Είναι μια πρόκληση, δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι μπορώ να χτίσω ιδιαίτερη σχέση μαζί σας. Όχι γιατί θα πρέπει να υλοποιήσουμε, εγώ πρέπει να υλοποιήσω μια υποχρέωση, όχι μόνο γι' αυτό, με, το, με την τυπική έννοια, αλλά γιατί και πολιτικό συμφέρον έχω γι' αυτό, αλλά και εσείς έχετε πολιτικό συμφέρον να ξεκινήσω μια συνεργασία τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορέσουμε τότε να δείξουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνε μας, όπως είπα πριν. Αυτό τι σημαίνει για μένα. Καταρχάς, να κάνω εγώ ό,τι πρέπει από πλευρά μου ή από πλευρά μα, που είναι πολύ περίπλοκο. Όχι μόνο στην γειτονία μα, αλλά και στην διευρυμένη γειτονία μα. Του γείτονε των γειτόνων μα. Ξεκινάω από τα Βαλκάνια. Η πολιτική διεύρυνση είναι όχι η καλύτερη, αν όχι η μόνη εγγύηση για, την, το μετασχηματισμό, τη δημοκρατία και την οικονομική ανάπτυξη. Προ Ανατολά. Χρειαζόμαστε και θα χρειαστούμε μεγαλύτερη προσοχή να δώσουμε στην περιοχή αυτή, να υποστηρίξουμε την Ουκρανία σε ό,τι αφορά την ασφάλειά της, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, πολιτική διαδικασία, οικονομικές προκλήσεις και ενέργεια, ενεργειακές προκλήσεις. Και θα πρέπει η Μολδαβία και η Γεωργία, ειδικά τους επόμενους μήνες, ε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει επίσης ε, να ασχοληθούμε με το Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον Ανατολικό γειτονά μας στη Ρωσία θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως την συμφωνία του ΜΙΣΚ, όλα τα σημεία, όλους τους τομείς και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για ειρήνη σε αυτή τη χώρα. Η Ρωσία, πριν από ένα μήνα ήμουνα εδώ και σας είπα ότι μπορεί να μην είναι εντέρος αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά είναι μια στρατηγική σημασία χώρα παγκόσμια και είναι και γείτονα για την Ουκρανία καταρχήν. Επομένως θα πρέπει να επανεξιολογήσουμε μαζί τις σχέσεις μας με τη Ρωσία τα επόμενα πέντε χρόνια. Είπα ότι χρειαζόμαστε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην Ανατολή και παράλληλα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και στον Νότο. Στην Μέση Ανατολή, ειδικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας αποτελεσματικός πληρωτής και θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικός παίκτη. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτύξουμε όλο και περισσότερο ένα κοινό πλαίσιο για κοινέ δράσει για να σταματήσουμε το Ισλαμικό κράτο, το ISIS. Δεν είναι κράτο. Δεν είναι το Ισλάμ. Αλλά είναι μια μείζωνα παγκόσμια απειλή που μα απειλεί όλου. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη, Λιδία, στη Λιβύη, που μπορεί να είναι επόμενη, ο επόμενο στόχο. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο μαζί με το ΝΟΙΕ και τι γειτονικέ χώρε. Αλλά θα πρέπει επίση να δώσουμε προσοχή και σε ιστορίες επιτυχίας. Να μην εγκαταλείψουμε και να μην ξεχάσουμε τις ε, ιστορίες αυτές ε, επιτυχίες που είναι η Τινησία και το Μαρόκο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά στον Νότο και στους νότιους γείτονες των νότιων γειτόνων μας. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουν απλώς ε, βοήθεια, αλλά να είναι και εταίροι πολιτικά. Και μια και με Ιταλίδα, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ορτικό κύκλο στα βόρεια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ήσυχο, σιωπηλό. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα μείνει σιωπηλό για πάντα ο βορρά αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην Ανατολή και στον Νότο. Και αυτό δεν είναι αντίφαση για μένα. Ξέρετε ότι οι κρίσει δεν περιμένουν τη σειρά του για να σκάσουν. Δεν μα περιμένουν. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να τα κάνουμε αυτά μαζί και να δραστηριοποιηθούμε σε όλα τα μέτωπα. Αλλιώ δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Ξέρω ότι είναι όλο και πιο δύσκολο. Και τελειώνοντα, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, τη δύσκολη εποχή, μπορούμε να βασιστούμε σε σημαντικού εταίρου που δεν είναι απλώ φίλοι μα, αλλά άνθρωποι με του οποίου μπορούμε να συνεργαστούμε, που είναι αξιόπιστοι. Η διατλαντική εταιρική σχέση, α πούμε, που είναι όλο και πιο στρατηγική και για την ασφάλεια, και είμαι έτοιμο να δουλέψω με τον Γιάνν Στότεμπερ, τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι καλός μου φίλος. Και οικονομικά, ξέρω ότι συζητάτε με τη Σεσίλια Τίτη. Και φαντάζομαι ότι κάποια ερώτηση θα μου γίνει γι' αυτό. Με τη Σεσίλια έχετε συζητήσει για το TTIP. Και τις παγκόσμιες απειλές. Επίσης, ε, άλλο στρατηγικός εταίρος είναι η Λατινική Αμερική όχι μόνο οι δύο στρατηγικοί εταίροι που έχουμε εκεί, αλλά η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική συνολικά είναι πιθανό στρατηγικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σύνοδο Κορυφή τη ΕΛΑΚ ε, έγινε τον Ιούνιο και είναι ε, μια τεράστια δυνατότητα για να επανεκκινήσει αυτή η σχέση. Είναι σημαντικό να μην του θεωρούμε δεδομένου. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολιτική δέσμευση εκεί από πλευρά μα. Μιλάω για την περιφερειοποίηση, που είναι μια αξία στην Λατινική Αμερική. Την έχω υπόψη μου. Και τώρα το μυαλό μου πάει στην Ασία. Εκεί θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, την Κίνια, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κορέα. Αλλά θα πρέπει επίσης να συνεργαστούμε και να λάβουμε υπόψη μας τις περιφερειακές ομάδες, τους περιφερειακούς σχηματισμούς ΑΣΕΝ και να συνεργαστούμε με αυτές. Και με χώρες οι οποίες δεν θεωρούμε κατά ανάγκη ότι είναι χώρες κλειδιά, αλλά όπου αν κάνουμε μια μικρή επένδυση μπορεί να δώσει πολλούς καρπούς. Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί με άλλες οργανώσεις περιφερειακές και παγκόσμιες. Ε, με τον ΟΗΕ προφανώς, ΝΑΤΟ, το ανέφερα, αλλά και περιφερειακές. Ο ΕΣΥ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, Αφρικανική Ένωση. Έχουμε και κοινή δουλειά να κάνουμε και κοινή ατζέντα για την ε, κλιματική αλλαγή που είναι τμήμα τη εξωτερική μα πολιτική και πρέπει να είναι όλο και περισσότερο στο μέλλον. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπου πιστεύω ότι ω Ευρωπαίοι έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να έχουμε μια συνεκτική ατζέντα και να συμπεριλάβουμε και τι εσωτερικέ μα πολιτικέ. Τρει βασικοί τομεί που θα ήθελα να αναφέρω. Ελευθερία των ΜΕ, γυναίκε και θρησκευτική ελευθερία. Τελευταίο και σημαντικό, και θα κλείσω με αυτό, η αναπτυξιακή ατζέντα του, 2015 ε, του, ΟΗΕ μετά το, 2015. Αυτό δεν αφορά μόνο τα κλασικά θέματα της ανάπτυξης, αλλά το περιβάλλον, την βιωσιμότητα και ταυτόχρονα ισχύει για την εξωτερική δράση και την εσωτερική δράση. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας.